So it's my pleasure to... Uh, Με χαρά καλωσορίζω σήμερα άλλη μία υπουργό της Προεδρίας της Φινλανδίας, ύστερα από τον Υπουργό των Αρμόδιο για θέματα γεωργίας και δασών. Είχαμε χθε την κυρία Υπουργό Γεωργίας. Σήμερα έχουμε την κυρία Μίκονεν Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και στη συνέχεια την Υπουργό Οικογενειακών Υποθέσεων και Κοινωνικών Υπηρεσιών, όπου βεβαίως θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ε, δημόσιας υγείας που ανήκουν στις αρμοδιότητες Επιτροπής μας. Και θα ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις κατόπιν της συνεδριάσεως των συντονιστών της 18 Ιουλίου. Πρέπει τυπικά για λόγους τυπικούς να ρωτήσω τους συντονιστές αν έχουν κάποιες παρατηρήσεις σχέση με τα πρακτικά που διενεμήθησαν ηλεκτρονικά. Δεν βλέπω παρατηρήσεις. Άρα μπορούμε να θεωρήσουμε πως έχουν εγκριθεί. Και μπορώ να σας ενημερώσω για δύο-τρία πράγματα από την ε, από τι αποφάσει που έλεγχαν στην πρώτη συνεδρία των συντονιστών. Η πρώτη απόφαση ήταν ε, να προσκληθεί η Επίτροπος Μάλστρομ στην πρώτη συνεδρία του Σεπτεμβρίου για το Mercosur ώστε να έχουμε το χρόνο να διατυπώσουμε ερωτήματα για την ε, εμπορική αυτή συμφωνία και τα θέματα των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας, δηλαδή κλιματική αλλαγή, ασφάλεια τροφίμων, βιοποικιλότητα. Θα αποσταλεί σήμερα η σχετική πρόσκληση. Άλλη μία ε, επιστολή, πρόσκληση θα αποσταλεί στην Επιτροπο στον Επιτροπο πάλι για συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Ε, με στόχο να ενημερωθούμε και να λάβουν απάντηση οι ερωτήσεις σας οι σχετικές με τις εξελίξεις της ε, στο πλαίσιο του περιορισμού, της συμφωνίας για τον περιορισμό των εκπομπών από την αεροπλοία, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να περιορίσει μακροπρόθεσμα εάν επεκταθεί το σύστημα ITS e ε, των δωρεάν ανταλλαγών και πιστοποιητικών ε, μεσοπρόθεσμα να περιορίσει τις αρμοδιότητές μας για παρέμβαση. Είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει, το έχουμε συζητήσει επί μακρόν και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι διεθνούς βέβαια εμβέλειας, παγκόσμιας εμβέλειας και πρέπει οπωσδήποτε να το συστήσουμε αφού θα επηρεάσει και τους εσωτερικούς μας ε, κανόνες. Περιμένουμε ε, να έρθει η Επιτροπή στην πρώτη αυτή συνεδρία του Σεπτεμβρίου. Και τελευταίο και τρίτο σημείο κοινή γεωργική πολιτική. Έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό με του τονιστέ και αποφασίσαμε να μην ξανανοίξουμε τη γνωμοδότηση, το θέμα τη γνωμοδότηση ΕΝΒ, αυτή που είχε κατατεθεί στο παρελθόν και ισχύει ακόμη, όπω την είχε υιοθετήσει η προηγούμενη σύσταση τη επιτροπή ΕΝΒ, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία, να μην ανοίξει δηλαδή σε συζήτηση όλο το πακέτο και σε μια επιστολή την οποία σήμερα θα αποστείλω στον ομολογό μου της Επιτροπής Γεωργίας. Προτείνω μια συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας πιθανών ε, συμβιβασμών. Ξέρετε ότι και η ΕΝΒΙ έχει αρμοδιότητες για το θέμα της μεταρρύθμισης της ανοθεώρησης της ΚΑΠ. Έχω δει δυσφορία να εκφράζεται από πολλούς και δει μέλη της Επιτροπής μας. Και έτσι λοιπόν θα προτείνουμε συζήτηση πιθανών ε, συμβαστικών τροπολογιών πριν να έρθει το θέμα στην Ολομέλεια. Αυτά σε επαφή με την Επιτροπή Γεωργίας και όπως είπα η επίσημη γνωμοδότηση όπως είχε, είναι η επίσημη απόφαση όπως αποφασίστηκε από τους συντονιστές θα αποσταλεί σήμερα στον Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας σήμερα το πρωί. Προβλέπεται δε ε, συνεδρία των συντονιστών της Άγκρη και από εκεί θα κριθεί η εξέλιξη της υπόθεσης λαμβανομένου βεβαίω υπόψη ότι η καθήλυνα αρμόδια είναι η άγκρη. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Τρία κύρια θέματα για τις ε, προσεχείς συνεδριάσεις. Ε, έχετε κυρία Υπουργέ τώρα το χρόνο, 10 με 12 λεπτά. Μα με συγχωρείτε, λησμόνισα κάτι ακόμα. Ως πρόεδρος της ΕΝΒ προσεκλήθην ε, στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Ίντα σήμερα που έχουν μια ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο Μάλστρομ για το θέμα της Μερκοσούρ. Συντονιστές και πρόεδρος της Ίντα μας προσκαλούν ε, μέσω του Πρόεδρου ε, με μια δυνατότητα να διατυπώσουμε και κάποιες ερωτήσεις συγκεκριμένες στην Επίτροπο και άρα θα χρειαστεί να φύγω από την συνεδρίασή μας και τη συζήτηση. Κάπου στις 10.30 θα επανέλθω όμως το ταχύτερο δυνατό και οπωσδήποτε είμαι βέβαιος ότι επάξια θα με εκπροσωπήσει ένας εκ των αντιπροέδρων στην ανταλλαγή απόψεων με εσάς κυρία Υπουργέ. Και ξανάρχομαι σε εσάς. Σας ευχαριστώ και πάλι που είστε εδώ, που είστε μαζί μας. Πολλές ερωτήσει, πολλές οι προσδοκίες για την Φιλανδική Προεδρία. Έχετε το λόγο για 10 με 12 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μαζί σας για να σας μιλήσω για την Φιλανδική Προεδρία. Και ξέρω ότι έχετε ήδη συναντηθεί με έναν Φιλανδό Υπουργό και μετά από μένα έρχεται κι άλλο ένας. Οπότε πολλά νέα από τη Φιλανδία, από εμά. Λοιπόν, τα σχέδιά μας της Φιλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου στον τομέα του περιβάλλοντος ε, και του κλίματος είναι η δικιά μου αρμοδιότητα. Και ας αρχίσουμε με τα δύσκολα στοιχεία. Ξέρετε ότι ο Ιούνιος του 2019 ήταν ο πιο ζεστός Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίω. Ο αριθμός αλλαγής παγκοσμίω όσον αφορά τη φύση τα τελευταία 50 χρόνια είναι κάτι χωρίς προηγούμενο στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτά είναι στοιχεία κλειδί που παίρνουμε από το Κοπέρνικος και από την έκθεση αξιολόγησης για την βιοπικιλότητα και το οικοσύστημα του IPBES. Τα μηνύματα επίσης από το IPCC για 1,5 βαθμό δείχνουν ότι η ευκαιρία να αποφύγουμε μία ανεπιστρεπτή ζημιά στο κλίμα και στην ανθρωπότητα περιορίζεται συνεχώς. Με άλλα λόγια δηλαδή πρέπει να αναλάβουμε δράση και να πάρουμε αποφάσεις τώρα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί με τους εαυτούς μας και με τους πολίτες μας. Έχουμε μια συστημική πρόκληση μπροστά μας και θα πρέπει από εκεί να ξεκινήσουμε για να εκπονήσουμε ευρωπαϊκές πολιτικές για τα επόμενα πέντε χρόνια. Έτσι λοιπόν, η Φιλανδία έχει αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε δύσκολους καιρούς και σε θεσμικές αλλαγές. Δύσκολη αλλά και κρίσιμη καιρή είναι αυτή. Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβουν τα πρώτα βήματά τους κατά τη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας και έχουμε σημειώσει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συζήτηση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την τώρα επιβεβαιωμένη Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από μια εβδομάδα θέλουμε μαζί να έχουμε ένα θετικό θεματολόγιο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε δύο προκλήσεις κλειδί των καιρών μας, που είναι η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βιοπικιλότητας. Τι σημαίνει όμως ένα τέτοιο θεματολόγιο για τους επόμενους έξι μήνες. Όσον αφορά το κλίμα και το περιβάλλον, η Φιλανδική Προεδρία θα έχει τρεις προτεραιότητες. Η πρώτη είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή, εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την κλιματική δράση. Δεύτερον, φιλόδοξο έργο για την βιοπικιλότητα μετά το 2020 και τρίτον, πρόθεση της κυκλικής οικονομίας. Πρώτον, λοιπόν, δράση για το κλίμα. Είναι προτεραιότητα για τη Φιλανδική Προεδρία να είμαστε στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την κλιματική δράση. Και ήδη έχουμε πολύ φιλόδοξους στόχους, τους πιο φιλόδοξους στόχους από όλες τις βιομηχανικές οικονομίες και δεσμευτική νομοθεσία μάλιστα που θα μας επιτρέψει να πετύχουμε τους στόχους μας και τις δεσμεύσεις μας. Όμως δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ γιατί για την Ευρωπαϊκή Ένωση το να είμαστε στην πρώτη γραμμή σημαίνει να δεσμευτούμε για κλιματική ουδετερότητα, όπως λέγεται, το 2050. Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε ώστε να πετύχουμε συμφωνία όσον αφορά τα κύρια στοιχεία της ε, μακροπρόθεσμης κλιματικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό πριν, πριν από τα τέλη της χρονιάς όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επίσης θα υπάρξουν διάφορες ανατομέα συζητήσεις στο Συμβούλιο για να προχωρήσουμε ε, στο έργο μας, να φροντίσουμε να υπάρχουν κίνητρα και οι συζητήσεις θα γίνουν σε διάφορα πλαίσια για τη μακροπρόχρονη δράση μας και στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής και Μεταφορών και Περιβάλλοντος, αλλά και άλλα σχήματα του Συμβουλίου και άτυπες συναντήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου θα συζητήσουν τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική ουδετερότητα. Επιπλέον έχουμε και τις προετοιμασίες για την ε, διάσκεψη της ε, γραμματείας του ΟΗΕ όσον αφορά την κλιματική δράση. Έτσι συναντηθήκαμε πριν από δύο εβδομάδες στο Ελσίνκι όπου και συζητήσαμε για το κοινό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάσκεψη αυτή. Αυτό που απεκόμισα εγώ από αυτή τη συζήτηση είναι ότι επιπλέον από το ότι θέλουμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα όσον αφορά τη δέσμευσή μας για την ολοκλήρωση της δικιάς μας μακροχρόνιας στρατηγικής, έχουμε και άλλα πράγματα σημαντικά να πούμε, ότι έχουμε ένα δεσμευτικό πλαίσιο για το 2030 και τις κλιματικές ε, πολιτικές τις εφαρμόζουμε σε διάφορες πολιτικές αλλά και στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να ανακοινώνει ή να ενημερώνει επίσης ε, τους ε, στόχους της όσον αφορά τις εθνικές συνεισφορές μέχρι το 2020. Έχουμε πολλές πολιτικές συζητήσεις που μας περιμένουν προκειμένου να ολοκληρωθεί το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τα τέλη της χρονιάς αυτής. Επίσης θα είμαστε και στην πρώτη γραμμή στην προετοιμασία της COP25 που θα γίνει στη Χιλή και για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που θα εγκριθούν στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Οκτωβρίου. Δεύτερη προτεραιότητά μας είναι η βιοπικιλότητα και αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε στην άτυπη συνάντηση Υπουργών για το Κλίμα και το Περιβάλλον. Τώρα θα συνεχίσουμε με το έργο που πρέπει να συνεχίσουμε και τις συζητήσεις που μας περιμένουν για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα στο Συμβούλιο το Δεκέμβριο. Η σκληρή αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε αρκετά πίσω από τους στόχους μας όσον αφορά τη βιοπικιλότητα, τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίω. Το πρόβλημα δεν είναι οι στόχοι μας, είναι η υλοποίηση των στόχων. Η απώλεια οικοτόπων, ε, πρακτικές που δεν είναι βιώσιμες, ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τη γη και το νερό μας, η υπερβολική χρήση των φυσικών όπορων αποτελούν σημαντικά στοιχεία του προβλήματος. Για μένα, ε, αυτό που αποκόμισα από τις συζητήσεις για τη βιοπικιλότητα είναι ότι υπάρχει ισχυρή βούληση για αξιόπιστα μέτρα και πλαίσιο, όπως επίσης και μετρήσιμη στόχη όσον αφορά την επόμενη δεκαετία. Αντιλαμβάνουμε επίσης ότι το να σταματήσουμε την απώλεια βιοπικιλότητας δεν έχει να κάνει μόνο με την προστασία της φύσης. Είναι κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλους τους ε, τομεκούς τομείς πολιτικής, όπως είναι και η κλιματική αλλαγή. Η Φιλανδική Προεδρία λοιπόν θα αρχίσει με φιλόδοξη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύμβαση για την Βιολογική βιοπικιλότητα και την διάσκεψη των μερών, το COP15 δηλαδή, που θα συμφωνήσει για στόχους μετά το 2020, τον Οκτώβριο του 2020, στο Kunming στην Κίνα. Στόχος της Φιλανδικής Προεδρίας είναι να βρει κοινό τόπο και να προετοιμάσει τις επόμενες διαπραγματεύσεις για την βιοπικιλότητα, όπως επίσης να συνεισφέρει και στο πλαίσιο για την βιοπικιλότητα μετά το 2020. Και έρχομαι στην τρίτη μας προτεραιότητα που είναι η κυκλική οικονομία. Η κυκλική οικονομία μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης στις ε, διτές ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και όσον αφορά το κλίμα και όσον αφορά την απόλυτη επικοινότητας. Αν περάσουμε στην κυκλική οικονομία θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και την κρίση βιωσιμότητα. Πρέπει λοιπόν να προσαρμόσουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την κυκλική οικονομία τον Οκτώβριο στο Συμβούλιο Περιβάλλοντο. Η κυκλική οικονομία συζητιέται επίση και στου υπουργού κλίματο και περιβάλλοντο και έγινε αυτό και στο Ελσίκη πριν από δύο εβδομάδε. Κυκλική οικονομία σημαίνει ότι διαχειριζόμαστε τα οικοσυστήματα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ανανεωθούν προκειμένου να διατηρηθούν οικολογικοί πόροι και να ανακάμπτουν οι φυσικές πηγές, ενώ βέβαια χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε και το κοινωνικό και οικονομικό παράγοντα που πλήττει τις τρέχουσες και τις επόμενες γενιές και το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς, η Προεδρία μας θέλει να βοηθήσει την Επιτροπή να έχει ένα ισχυρό μήνυμα όσον αφορά την κυκλική οικονομία και για τα επόμενα πέντε χρόνια. Σε πολλούς τομείς, όπως είναι ο οικοδομικός τομέας, η φαντουργία, η... ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σπαταλούνται πάρα πολλοί πόροι. Με τις κατάλληλες πολιτικές όμως και τις κατάλληλες προδιαγραφές μπορούμε να επιτρέψουμε στις πρώτες ύλες να κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή οικονομία και να παράγουν αξία θα πρέπει να σχεδιάζονται τα προϊόντα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πιο εύκολο να επισκευαστούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν. Η κυκλική οικονομία περιορίζει την ανάγκη για καινούριε πρώτε ύλε και μειώνει και τι εκπομπέ και γενικά την ε, πίεση πάνω στο περιβάλλον. Επιπλέον, η ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή οικονομία θα βασίζεται σε πιο αποτελεσματικέ και πιο βιώσιμε ε, πρώτε ύλε κυκλική οικονομία έχει νόημα ανεξάρτητα από ποια οπτική γωνία το κοιτάει κανεί. Η επιτυχία λοιπόν αυτών των τριών προτεραιοτήτων μα και τη πολιτική μα γενικότερα βασίζεται και στην καλή υλοποίηση. Εδώ έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία στη διάθεσή μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα προγράμματα που σίγουρα έχουν επιπτώσει θετικέ όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον είναι το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για το περιβάλλον, το οποίο ε, καταθέτει μία ε, σημαντική στρατηγική και δημιουργεί συσχετισμούς με θετικά μέτρα. Το έβδομο αυτό πρόγραμμα επίσης έχει συνεισφέρει σε καλύτερο και πιο γρήγορο συντονισμό στον τομέα του περιβάλλοντος και της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή. Επιτρέπει επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκφράζεται με μία φωνή στο διεθνές πλαίσιο και στις διαπραγματεύσεις που γίνονται εκεί. Το 7ο λοιπόν ε, πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον μέχρι τα τέλη της επόμενης ε, χρονιάς ε, θα έχει ολοκληρωθεί, αλλά χρειάζονται παρετέρω δράσεις. Και γι' αυτό το λόγο η Φιλανδική Προεδρία έχει ως στόχο να προσαρμόσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου όσο γίνεται καλύτερα προκειμένου να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο για το περιβάλλον και να βασιστεί βέβαια στα επιτεύγματα και τις επιτυχίες του 7ου και να διασφαλίσει την συνέχεια του στρατηγικού πλαισίου για το κλίμα και τις δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος. Ας δούμε λίγο τώρα και τους νομοθετικούς φακέλους, τους οποίους θα επεξεργαστεί η Φιλανδική Προεδρία. Έχουμε δύο που σχετίζονται με το πόσιμο είδωρ και την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. Στόχος λοιπόν της Φιλανδικής Προεδρίας είναι να αρχίσει και να ολοκληρώσει του τριμερεί διαλόγους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την Προεδρία μας. Επίσης, όσον αφορά το MRV. Επίσης, στόχος μας ε, είναι να προχωρήσουν οι θέσεις του Συμβουλίου και να ολοκληρωθούν στην Προεδρία μας. Για το LIFE, επίσης, έχουμε διαπραγματεύσεις και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί και αυτός ο φάκελος που σχετίζεται βέβαια και με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Επιτροπή σας και το έργο σας, να ξέρετε ότι πάντα ήταν βασικό για μας και θα συνεχίσει και τα επόμενα πέντε χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα θετικό θεματολόγιο και να δώσουμε απαντήσεις στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας σε σχέση με το κλίμα και την απώλεια βιοπικιλότητας. Τώρα, κοιτώντα την γενικότερη εικόνα, η κοινή γεωργική πολιτική μαζί με ε, βιώσιμα δημοσιονομικά είναι δύο ε, σημαντικοί παράγοντες για την αλλαγή που χρειαζόμαστε και τη μετάβαση που χρειαζόμαστε. Και ακόμα και αν το, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος δεν είναι υπεύθυνο για αυτές τις πολιτικές από πλευρά του Συμβουλίου, οι συζητήσεις αυτές θα προχωρήσουν όμως στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλίας, αλλά και στο Συμβούλιο Οικονομικών Υποθέσεων. Χρειαζόμαστε μία προσέγγιση ολοκληρωμένη και διατομιακή αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Να ενσωματώσουμε καλύτερα τις πολιτικές μας για το κλίμα και το περιβάλλον σε άλλες πολιτικές, ξεκινώντας βέβαια από το καθημερινό μας έργο. Και γι' αυτό και η υλοποίηση του θεματολογίου 2030 για την βιώσιμη ανάπτυξη τόσο παγκοσμίω όσο και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας. Και έτσι έρχομαι πάλι στη διεθνή σκηνή. Έτσι ξεκίνησε και την ομιλία μου. Έχουμε πετύχει πολλά τα τελευταία χρόνια όσον αφορά το κλίμα και το περιβάλλον και όσον αφορά τους ε, βιώσιμους στόχους μας, τόσο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσμίω. Όμως η επιστήμη είναι ξεκάθαρη, όπως είναι και αυτά που ζητάει η κοινωνία των πολιτών, η οποία φωνάζει όλο και πιο δυνατά και λέει ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και ότι πρέπει να αρχίσουμε τώρα, αμέσως. Το παράθυρο ευκαιρίας που έχουμε μπροστά μας κλείνει όλο και περισσότερο και γρήγορα. Αλλά θέλω να τελειώσω με μια πιο αισιόδοξη νότα, ότι παραμένει ένα παράθυρο ευκαιρία μπροστά μα, ένα ανοιχτό παράθυρο. Και έχουμε πολύ σημαντικέ πολιτικέ αποφάσει να πάρουμε. Αγαπητά μέλη τη Επιτροπή Περιβάλλοντο, σα εύχομαι αφοσίωση, σοφία και πάθο όταν φέρετε σε πέρα στο έργο σα τα επόμενα πέντε χρόνια. Προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας για να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις των καιρών μας. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας υπενθυμίσω ότι οι συντονιστές θα έχουν στη διάθεσή τους έκαστος δύο λεπτά για τις ερωτήσεις τους. Αυτός θα είναι ο πρώτος γύρος με 7 συγκεκριμένα ερωτήσεις. Θα έχετε, κυρία Υπουργέ, στη διάθεσή σας 7 με 10 λεπτά να απαντήσετε και θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος ερωτήσεων από τους ευρωβουλευτές. Σας ενημερώνω επίσης πως ε, ακυρώθηκε η πτήση της Εσίλια Μάλστρομ, άρα το μεσημέρι θα γίνει ακρόαση, που σημαίνει ότι εγώ θα συνεχίσω να προεδρεύω. Συγγνώμη, Μπάς, δεν ξέρω αν είναι εδώ. Έφυγε ήδη. Α, όχι, εδώ είναι. Εδώ είναι. Ναι, τώρα μπορείς να κοιμηθείς ήσυχο. Να ξεκινήσουμε τον Πέτερ Λίζε από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Η, ε, πρόεδρος, η νέα πρόεδρος Κομισιόν έβαλε στο κέντρο της ομιλίας της την προηγούμενη τρίτη στο Στρασβούργο το κλίμα και μας ανέφερε πολύ φιλόδοξους στόχους ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προτάσεις. Ε, κάτι το οποίο χαιρετίζω ιδιαίτερα είναι το γεγονός ε, πως ε, σε ό,τι αφορά τις εναέριες μεταφορές, τις αεροπορικές μεταφορές ε, δήλωσε ότι θα αναλάβει δράση. Υπάρχει μια πραγματικά παράλογη κατάσταση ότι δεν χρησιμοποιούνται παρκώς οι σιδεδρομικές μεταφορές που θα μπορούσαν να μειώσουν την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από τις εκπομπές και αυτό είναι κάτι άλλο που το απαιτούν από εμάς οι πολίτες και ελπίζω να στηρίξουμε τα σχέδια της Φοντερ σε ό,τι αφορά τις ενέργειες μεταφορές. Ένα άλλο επίγον ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει είναι ότι η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αγορής και αναφέρθηκε αυτό προβλέπει μια συμφωνία ε, που θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην ε, ε, ανταλλαγή δικαιωματοπόδου και θα δημιουργήσει πρόβλημα με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, ώστε να στηριχθούν τα κράτη που εξαρτώνται από τον άνθρακα ακόμη. Χρειάζεται βέβαια γι' αυτό χρηματοδότηση και ο Πρωθυπουργό και άλλοι ε, δεν έχουν ακόμη αποφασίσει τι θα γίνει με αυτό το θέμα, ενώ έχουμε πολλέ νέε προκλήσει να αντιμετωπίζουμε. Νομίζω ότι καλό είναι όμω να έχουμε επαρκεί πόρου για τι σημαντικέ αυτέ προκλήσει. Επίση, η ε, προστασία του κλίματο είναι μια παγκόσμια πρόκληση. Βλέπουμε όμω κάποια βιομηχανικά κράτη, η ΙΠΑ αλλά και η Ιαπωνία, Αυστραλία και πολλέ άλλε που ε, σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες που κάνουμε εμείς ε, με τις ε, για την επίτευξη των στόχων των Παρισίων ε, δεν ε, έχουν και αυτές ακόμη καταλήψει στις δράσεις τους και θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση σε παγκόσμιο επίπεδο γιατί πρόκειται για παγκόσμιο ζήτημα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο ΣΕΠ Ντάνς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ που μας ε, παρουσιάσατε σε ποιους τομείς ε, θα εστιάσετε και κάποια ε, νομοθεσία που ακόμη κρέμει αναφέρατε. αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι ότι σε σχέση με την ανάγκη να εστιάσουμε στο πώς οι άνθρωποι αντιδρούν στην κλιματική αλλαγή και δεν ξέρω κατά πόσον εμείς ε, ε, είμαστε στο επίπεδο των προσδοκιών των πολιτών ε, που είναι έτοιμοι να κάνουν περισσότερα σε προσωπικό επίπεδο και το αν ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες με την νομοθεσία που θέλουμε να καταθέσουμε. Θα ήθελα να αναφέρω ε, την ε, διαμαρτυρία των κίτρων γυλαίκων στη Γαλλία με τους ενεργειακούς φόρους ε, που αυτό θεωρήθηκε λανθασμένα όμως αν επίθεση βάρος της καθημερινότητας, της καθημερινής ζωής των πολιτών. Και ο τρόπος το τον πολίτες πρέπει να ληφθεί υπόψη από εμάς. Δεν ξέρω αν προβληματίζεται καθόλου από αυτού δηλαδή η κυβέρνηση, δηλαδή για το πώς μπορεί να συνεργαστεί με Συμβούλιο και τα κράτη για να γίνει αυτή η αλλαγή ε, παραδείγματος. Διότι τι παρακολουθούμε. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα για το οποίο μιλήσατε και είπατε ότι ε, συρρυκνώνεται και θα συρρυκνωθεί και ακόμη περισσότερο Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι στις δράσεις μας. Όσο πιο φιλόδοξες θα είναι όμως οι δράσεις που θέλουμε να φέρουμε σε πέρα, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η αντίδραση. Εσείς πώς θα προωθήσετε αυτήν την άλλη παραδείγματος. Έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις, παραδείγματος χάρη, ε, και κονδύλια για μια δίκαιη μετάβαση ώστε να υπάρξει η χρηματοοικονομική υποστήριξη προς όσους είναι στην αιχμή ε, της τεχνολογίας και της πρόοδου προς, αυτό. Δεν ξέρω αν είχατε συζητήσεις και αν είχατε ή είδατε κάποια προθυμία από τα άλλα κράτη-μέλη για να γίνει συλλογικά αυτό το έργο. Διότι πρέπει να γίνει πραγματικά πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολύ σύντομα. Thank you, ευχαριστώ, Νίλ Στόρβαλς, για το Renew. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και να καλωσορίσω την Υπουργό στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είπατε στην ομιλία σας ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερο Και είμαι βέβαιο ότι όλοι μα το αντιλαμβανόμαστε και οι πολίτε επίση το συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο και στις αρχές του αιώνα και τη δεκαετία αυτή, οι στόχοι δεν ήταν ίσω όσο φιλόδοξοι θα μπορούσαν να είναι. Γιατί αν ήταν θα μπορούσαμε να του είχαμε επιτύχει και σε πρόστα. Το πρόβλημα είναι όμως ότι είναι πολύπλοκο το ζήτημα και συζητάμε διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος. Βλέπουμε δε ότι οι διάφοροι συμβαλόμενοι, οι διάφορες ΜΚΟ και άλλοι ξεκινούν από διαφορετικά σημεία κίνησης και από άλλη οπτική γωνία τα βλέπουν τα πράγματα ο καθένας. Έχουμε το στρατηγικό έγγραφο της Κομισιόν ο στόχος της νομίζω με αυτό ήταν να δημιουργήσει ένα σύστημα όπου τα κράτη-μέλη θα ορίζουν πώς αυτά θα προχωρούν ατομικά το καθένα σε ένα ουδέτερο ως προς το κλίμα μέλλον. Όμως η κατάσταση μας δείχνει πόσο μεγάλη ε, ιδιαιτερότητα χαρακτηρίζει το κάθε κράτος, άρα δεν μπορούμε να έχουμε one size fits all, ένα μέγεθος για όλους, ίδια πράγματα για όλους. Καλό θα ήταν και ενδιαφέρον θα ήταν να ακούσω εσείς τι πρεσβεύετε. Πώς να το πω, για αυτό το πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Πώς ξεκινάμε, από πού ξεκινάμε. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, ε, my... Ευχαριστώ. Μιχαήλ Μπλος, πράσινη. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ κύριε Υπουργέ Ξεκινώ χαίροντα σας για το σχέδιο για την προβολή της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης θερμοκρασίας του πλανήτη, για την πρωταγωνιστική δράση που οδηγεί σε μια ουδέτερη κλιματικά Φιλανδία στο το 2035. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι έχω μιλήσει με πολλούς νέους και με πολλούς νέους συναδέλφους εδώ στο Κοινοβούλιο Φοβούμαστε λοιπόν ότι το μέλλον διαμορφώνεται υπό και από την κλιματική κρίση. Βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο καμπής, πιστεύω όλοι συμφωνούμε, σε ένα σημείο που πλέον δεν θα μπορεί να ανατραπεί ή να αναστραφεί η κλιματική αλλαγή και η αύξηση θερμοκρασία του πλανήτη, εάν δεν αναλάβουμε αμέσω δράση. Πρέπει λοιπόν και φέρουμε εμεί την ευθύνη να δείξουμε την υπευθυνότητα και τη φιλοδοξία που χρειάζεται. Χθε ε, ο Γενικό Γραμματέα ζήτησε μία πρόταση για αύξηση, για μείωση γνώμη των ε, ρήπων στον Αύγουστο. Ε, τι θα πείτε εσείς ως Συμβούλιο στο Γενικό σας Γραμματέα, θα το Γενικό Γραμματέα των Εθνών. Θα δεσμευθείτε ε, για τον στόχο του 1,5 βαθμών. Επίσης, για τη χιλή, πάλι πρέπει να δώσουμε, να δώσουμε δείγματα φιλοδοξίας και πολλά είναι αυτά τα οποία έχουμε να κάνουμε όταν μιλούμε για στόχους έως και 40%. Ε, που δεν είναι συμφωνό όμω με το Παρίσι, με τι απαιτήσει του Κοινοβουλίου και τις φιλοδοξίες ε, των πολιτών που πήγαν στην κάλπη στι ευρωεκλογέ. Πώς λοιπόν θα μπορέσετε να ξαναβάλλετε στην πρώτη γραμμή της πρωτοπορία στην Ευρώπη και να επιδιώξετε το στόχο του, της κατά 50% έως το 2030. Επίσης, πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως, είπατε. Ναι. Η κλιματική αυτή κρίση Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να λυθεί μόνο με το να κλείνουμε τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες ε, το βράδυ, γιατί αυτό είναι το πιο εύκολο και το πιο ε, ανέξοδο ε, μέτρο. Τι άλλο έχετε να προτείνετε. Ευχαριστώ πολύ, Ελκονάινεν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ. Το κλίμα πάντα άλλαζε σε όλη την ιστορία του πλανήτη. Αλλάζει το κλίμα και θα εξακολουθεί να αλλάζει. Ακόμα και σε μια εποχή των παγετών μπορεί να ξαναγυρίσουμε και βέβαια καθοριστικό ρόλο έχει ο ήλιος. Ο ήλιος καθορίζει τι συμβαίνει στον πλανήτη μας βράχει πρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Έτσι λοιπόν, δεν έχουμε απεριόριστα μέσα για να αντιμετωπίσουμε την εξέλιξη. Τώρα βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή έχει μετατραπεί σε μια νέα θρησκεία και είναι βλασφημία και το να την αναμφισβητήσει κανείς. Κάποιοι μιλούν για αύξηση θερμοκρασία του πλανήτη, αλλά οι μακροχρόνιε στατιστικέ δεν την αποδεικνύουν ως φαινόμενο. Είναι ψευδείς αυτές οι στατιστικές που στηρίζουν τον ισχυρισμό της μακροπρόθεσμης αύξησης της ε, θερμοκρασίας του πλανήτη, ο οποίος είναι μια χαρά στην υγεία του, σας διαβεβαιώ. Ε, μας προξενεί μεγάλη δυσφορία το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Φιλανδίας έχει πέσει μέσα σε αυτήν την ε, παγίδα και προσπαθεί να εισαγάγει μέτρα με νέα φορολογία και τα λοιπά που θεωρείτε ότι είναι καλά. Στο παρελθόν η Εκκλησία πουλούσε όπλα. Ε, τώρα βλέπουμε να το ξανακάνει αυτό όταν ζητάει το παγκάρι να πάει να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Λοιπόν, έχουμε κάποια αποφάσει. δεν θυμάμαι καν τα νούμερα και, τα, και τους ορισμούς που έχετε πάρει για τις εκπομπές, αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι χώρε ε, αναπτυσσόμενε όπω η Ινδία και η Κίνα που έχουν εκπομπέ 30 κονταπλάσιε από τι εκπομπέ των ευρωπαϊκών κρατών, δεν πρέπει αυτέ να τι κρίνουμε πιο αυστηρά. Αυτέ τι χώρε pigs όπω τι λέμε. Ευχαριστώ, επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία, πολύ καλή επιτυχία στο έργο σας. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. κλιματική αλλαγή και Green Deal. Ναι, πολύ καλό να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα μαζί, αλλά μόνο εάν φέρουν αποτελέσματα οι νομοθεσίες, ε, τα νομοθετήματα που εισάγουμε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και αυτό βέβαια είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα και ερωτήματά μου. Είστε διατεθειμένοι να επιχειρήσετε να πείσετε τους εταίρους εκτός Ευρώπης να ακολουθήσουν αυτές τις τάσεις. Και δεύτερον, θα επηρεάσουν ε, εις βάθος βέβαια το, τη βιομηχανική μας παραγωγή, τις κοινωνίες μας, την, ε, παραγωγή την ε, οικονομία μας. Το είδαμε με την αντίδραση των πολιτών όταν έγινε μια προσπάθεια για επιβολή φόρου διοξιδίου του άνθρακα. Άλλωστε δεν έχουν όλες οι κοινωνίες την ίδια ε, διάρθρωση τη οικονομία του. Η, η Πολωνία Φερρυπίν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα ε, για την οικονομία της. Σε αυτό το βαθμό λοιπόν, τι μπορείτε να κάνετε και πού θα βρείτε τα χρήματα για να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Από τις παρατηρήσεις μου τα τελευταία χρόνια διαπιστώνω ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει ως κύριο πρόβλημα όχι τόσο την αύξηση θερμοκρασίας όσο την ξηρασία και βέβαια νομίζω ότι πολύ σωστά επισημαίνεται ως πρόβλημα η εκρίζωση των δασών και η αποψήλωσή του στην Αμαζο... στον Αμαζόνιο και την Ινδονησία, αλλά στην Ευρώπη έχει τεράστιο ε, τεράστια συνέπειες επίσης η αποψηλώση των δασών και γι' αυτό δεν γίνεται λόγος όπως δεν γίνεται και λόγος για το νερό σαν μέσον, σαν μάλλον ανάγκη διαφύλαξης των ε, υδάτινων πόρων στην Ήπεθρο και καταπολέμησης της ξηρασίας που θα έχει τεράστιες συνέπειες για τους πολίτες αλλά και τη βιοπικιλότητα. Αυτό ήταν η ερώτησή μου, αφορούσε δηλαδή τη διαχείριση των υδάτων. Τελευταίος, εκ τελευταία εκ μέρους των στολιστών, κυρία Μόντι Γκουέ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μίκοναν, είναι δύσκολη η εποχή που αναλαμβάνετε την Προεδρία, μεγάλες οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και ιδιαίτερα σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την ε, εστίαση ως προτεραιότητα στην κλιματική αλλαγή στο πρόγραμμά σας. Ε, θα ήμασταν παλαβή βέβαια να αμφισβητούσαμε την κλιματική αλλαγή όταν υπάρχουν ε, επιστημονικά στοιχεία και όταν υπάρχουν και επιστημονικέ λύσει στο πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ η Φινλανδία πώ μπορεί να προαγάγει την ιδέα ότι η οικολογική αναδιάρθρωση μπορεί να γίνει με τρόπο και κοινωνικά ε, δίκαιο και ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες ε, των πολιτών και βεβαίως αναλόγως και των διαφορετικών τους ε, οικονομικών δυνατοτήτων και εισοδημάτων. Η Φινλανδία στο το 2050 θέλει να είναι ουδέτερη ως προς τον άνθρακα, ε, ωστόσο νομίζω ότι μπορούμε και να έχουμε ταχύτερες λύσεις όπως μείωση ως το 2030 κατά 55% των εκπομπών. Το σύστημα ανταλλαγών, ETS πρέπει επίσης να εξελιχθεί περισσότερο. Ε, είδαμε συζήτηση να γίνεται και από άλλου υπουργού και για τις δεξαμενές άνθρακα, αλλά για, την, για την αποψήλωση των δασών δεν ε, συζητούμε επαρκώς. Ε, εσείς λοιπόν τι έχετε να προτείνετε, έχετε κάποια μέτρα που μπορούν να δώσουν κατευθύνσεις, είπατε κι εσείς ότι καθυστερούμε σε σχέση με την, με την καταπολέμηση της απώλειας βιοπικιλότητας και βέβαια η βιοπικιλότητα από μόνη της είναι απαραίτητη, είναι μια αυταξία. Ωστόσο πρέπει ταυτόχρονα και να κοιτάξουμε ε, την συμβολή της στην κλιματική αλλαγή και το βαθμό μέσα στον οποίο μπορεί να συμβάλλει. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε ώστε ε, μέσα στην Φιλανδική Προεδρία να αλλάξουμε κατευθύνσεις και να διαφυλάξουμε τη βιοπικιλότητα και για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής. Oh, ευχαριστώ, ναι. Ευχαριστώ για τον πρώτο γύρο. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας, παρακαλώ, για να απαντήσετε σε αυτό τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ και θα μιλήσω φιλανδικά τώρα, οπότε αν θέλετε να καταλάβετε, βάλτε τα ακουστικά σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις τόσο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Άκουσα πολύ καλές παρατηρήσεις ε, σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε μαζί από κοινού προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Ένα πρώτο θέμα που άκουσα είναι ότι πρόκειται για μια δράση βραχυπρόθεσμη που πρέπει να αναλάβουμε ε, δεν ε, φτάνει δηλαδή να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα, πρέπει και βραχυπρόθεσμα να κάνουμε κάτι. Ο Πίτερ Λίζε αναφέρθηκε σε φιλόδοξους ε, στόχους της κυρίας Φοντερ Λάιεν. Ναι, το κοιτάξαμε και αυτό και ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ που τόνισε διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και το κλίμα και η Φιλανδική Προεδρία θα έχει πολύ παρόμοιους στόχους. Άλλο εκπρόσωπος του Συμβουλίου καταλαβαίνετε ότι εγώ θα πάω πάρα πολύ σε βάθος για να πιέσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δουλέψει πάνω σε αυτά. Πάντως χαίρομαι που ακούστηκαν όλα αυτά που είπατε. Και είναι αλήθεια ότι μας περιμένει σκληρή δουλειά για να πείσουμε και άλλες χώρες. Και έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε και μπορούμε να το κάνουμε. Ε, μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας, αλλά θα πρέπει και οι άλλες χώρες να συνεισφέρουν, να πιστούν και άλλες χώρες να μας ακολουθήσουν σε αυτό. Ο κόσμος λέει ότι θέλει να κάνει περισσότερα από τη μια, από την άλλη μεριά αντιστέκεται κάθε φορά που λαμβάνονται αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις δύο τάσεις. Ξέρουμε ότι οι νέοι ανησυχούν πάρα πολύ για το μέλλον τους και αυτό έχει φανεί ξανά και ξανά και το ακούμε από τους νέους ότι θέλουν συγκεκριμένη δράση. Συγχρόνως όμως γνωρίζουμε ότι όταν λαμβάνουμε αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα του πολίτη, υπάρχει μια ομάδα πολιτών που αντιδράει. Και το είδαμε αυτό με διάφορα κινήματα που δημιουργήθηκαν. Είναι πολύ σημαντικό να προτείνουμε λύσεις οι οποίες να είναι και κοινωνικά βιώσιμες. Σίγουρα δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό και καταλαβαίνουμε ότι έχουμε διαφορές μεταξύ μας ε, ιστορικά, επειδή έχουμε επιλέξει διαφορετικές ενεργειακές λύσεις ο καθένας στη χώρα του. Αλλά όλοι θέλουμε να απαλλαγούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Συγχρόνως όμως πρέπει από κοινού να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις που να ταιριάζουν σε ολόκληρη την Ευρώπη προκειμένου η Ευρώπη να πετύχει τους στόχους της. Πρέπει να μειώσουμε την κλιματική αλλαγή. Άρα χρειάζεται δουλειά ανατομέα. Ε, με ρωτήσατε από πού να ξεκινήσουμε. Δεν υπάρχει ένα μόνο τομέας. Όλοι οι τομείς και όλοι οι κλάδοι επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή. Άρα το τι θα κάνουμε ε, δεν θα είναι σε ένα μόνο τομέα, σε πολλούς δράσεις για το κλίμα, την ενέργεια, τις μεταφορές, τον οικοδομικό κλάδο. Ολόκληρη η ανθρώπινη δράση, κάθε τομέα της πρέπει να αλλάξει. Γιατί μόνο έτσι θα καταλήξουμε σε λύσεις που να είναι καλές για το περιβάλλον. Τώρα, ε, Επιστήσατε επίσης την προσοχή μου στην διάσκεψη του ΟΗΕ. Φυσικά και θέλουμε την ε, ουδετερότητα όσον αφορά τον άνθρακα. Από την άλλη μεριά ε, θα πρέπει να είμαστε συμβατοί με ό,τι λέει η Συμφωνία των Παρισίων. Και στόχος της Φιλανδικής Προεδρίας είναι να το κάνουμε αυτό, να τηρήσουμε δηλαδή τις υποχρεώσεις μας. Όλοι στην Ευρώπη πρέπει να σκεφτούν πρακτικές λύσεις και να διασφαλίσουμε ότι οι δράσεις μας ευθυγραμμίζονται πάντα με τη Συμφωνία των Παρισίων. Πάνω σε αυτό πρέπει να συζητήσουμε παραπάνω. Ο κύριος Χάκενάιν δίστασε και αμφιβάλλει για την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής, κατά πόσο είναι πραγματική όχι, γιατί λέει ότι ήταν πάντα μια μεταβλητή. Πράγματι υπήρχαν μεταβολές στο κλίμα, υπήρξαν ε, εποχές παγετώνων, όλα αυτά, ναι, πράγματι. Αλλά είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι η κλιματική αλλαγή υπάρχει και οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία αν μη τι άλλο επιτάχυνε τη διαδικασία αυτή. Συνεπώς πρέπει να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και υπάρχει συνένεση στον επιστημονικό κόσμο επ' αυτού, ότι υπάρχει δηλαδή κλιματική αλλαγή και ότι είναι ανθρωπογενής. Δεν θα απαντήσω σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τη Φιλανδία, γιατί εδώ εκπροσωπώ το Συμβούλιο συνολικά και όχι μόνο τη Φιλανδία. Ο κύριος Βόντου. είπε ότι πρέπει εμείς να είμαστε το παράδειγμα και τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να πείσουμε και άλλες χώρες να μας ακολουθήσουν. Αυτά που κάνουμε εμείς είναι ένα μήνυμα για τους άλλους έτσι κι αλλιώς. Έχουμε know-how στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε δυνατότητες τεχνολογικές έχουμε την ε, δύναμη των δημοκρατιών μας. Δεδομένων λοιπόν όλων αυτών, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι χώρες της δεν δίνουν καλό παράδειγμα, σαφώς και θα ήταν πάρα πολύ περίεργο αυτό και θα ήταν ε, δύσκολο να πείσουμε τότε και άλλους να ακολουθήσουν το καλό παράδειγμα. Πρέπει λοιπόν να κοιτάμε μακροπρόθεσμα, αλλά ακόμα και βραχυπρόθεσμα. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε πάνω σε αυτό τον πλανήτη, πώς θα συνεχίσουν να είναι ζωντανές οι κοινωνίες μας. Υπάρχει και αλληλοεξάρτηση εξάλλου. Και όπως έχω ήδη πει, η κάθε χώρα έχει τη δικιά της ιστορία και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Και να καταλήγουμε σε λύσεις για αλλαγέ, συγχρόνως στηρίζοντας τις περιφέρειες. Έχουμε το know-how στην Ευρώπη, όπως είπα, μπορούμε να βοηθήσουμε ε, σε κατάρτιση τον κόσμο στις περιφέρειες εκείνες που βρίσκονται πιο πίσω, που κινδυνεύουν περισσότερο από τα μέτρα για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής κλπ. Και θέλουμε να έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ξηρασία, την ανιδρία που οφείλονται στο ε, αύξηση βέβαια της θερμοκρασίας, στην ε, μεγάλη ζέστη. Η διαχείριση των υδάτων είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι της ε, πολιτικής μας επίσης. και ε, στοχεύουμε σε μια συμφωνία η οποία θα καλύπτει το θέμα της επανάχρησης των υδάτων. Επίσης, θέλουμε να βρούμε ασφαλείς τρόπους επανάχρησης των υδάτων ε, και, σε αυτό, και αυτό εντάσσεται και στην ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους υδάτινους πόρους. Επίσης, η κοινωνική δικαιοσύνη που αναφέρθηκε. Ναι, είναι κρίσιμο θέμα. Οι διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να προχωρήσουν κατά τρόπο οργανωμένο και δίκαιο για να είναι και αποδεκτές. Θέλουν οι πολίτε να κάνουν περισσότερα, αλλά πρέπει να κατανοούν και αυτό που κάνουμε και να είναι ε, δίκαιες κοινωνικά οι συνέπειες ή τα μέτρα που θα εισάγουμε για να επιτύχουν. Η βιοπικιλότητα. βιοπικιλότητα όντω έχει κάπω επισκιαστεί από τον κίνδυνο τη κλιματική αλλαγή, παρότι υπάρχει σαφή διασύνδεσμο μεταξύ του. Γιατί και η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε απώλεια βιοπικιλότητα και ξέρουμε πολύ καλά ότι όσο περισσότερη είναι η βιοπικιλότητα, τόσο και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα τη φύσης και η προσαρμοστικότητά της. Και γι' αυτό έχουμε και το στόχο της ενεργοποίησης της συμφωνία για τη Βιοπικιλότητα το ταχύτερο δυνατό, ώστε να φέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και αυτό βέβαια ε, να σημαίνει να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση και με άλλες χώρες. Μπορούμε να έχουμε μια καλή συνθήκη. Είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό. Πρόοδο δεν έχουμε δει ε, στην πράξη, αλλά πιστεύω ότι όσο, είναι, όσο καλύτερα είναι τα μέτρα που εισάγουμε, τόσο πιο σωστή και η υλοποίησή τους. Και βεβαίως η υλοποίηση έχει κρίσιμο χαρακτήρα. Αυτό το βλέπουμε και στη συνθήκη των Παρισίων που έχει υποδειγματικό χαρακτήρα για το πώ θέλουμε να προχωρήσουμε. Δηλαδή θέλουμε σαφείς στόχου, σχέδια αναχώρα, σαφείς δεσμεύσεις, σαφείς υποχρεώσεις, μετρήσιμους στόχου και μέτρηση των, ε, του βαθμού επίτευξή του φυσικά. Αυτά, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προχωρήσουμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Επτά για τον πρώτο γύρο. Θα σας δώσω πέντε με επτά λεπτά, κύριε Υπουργέ, εν συνεχεία να απαντήσετε και θα ακολουθήσει επόμενος γύρος. Εντίνα Τόφ από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλήσατε την κλιματική προστασία Ω μία από τι βασικές προτεραιότητες της φιλανδική Προεδρίας. Διότι πραγματικά πρέπει να καθοριστούν και να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι κατά τρόπον ώστε να μην πλήξει αυτό την ανταγωνιστικότητά μας και να μην ε, οδηγηθούν όμως ε, τρίτες χώρες να αυξήσουν τις εκπομπές τους. Ε, η ουδετερότητα προ τον άνθρακα είναι μια, μια στρατηγική. Απαιτεί περισσότερη συζήτηση, όχι όμω ιδεολογικού χαρακτήρα. Κατά την άποψή μου, πρέπει να εστιάσουμε στι αναλύσει. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αγωνίζονται και αυτά για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Οι κλιματικοί στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν με τρόπο τεχνολογικά ουδέτερο. Να υπάρχει επαρκή προπολογισμό από ενωσιακή πλευρά για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων. Και είναι σημαντικό όλε τι πλευρέ να συνεισφέρουν στην υλοποίηση τη Συμφωνία των Παρισίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το καλό παράδειγμα, ωστόσο πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες χώρες ε, από τον υπόλοιπο κόσμο, να θέσουν και αυτές οι χώρες φιλόδοξους στόχους. Αγαπητοί Υπουργέ, ποιοι είναι οι στόχοι της Φιλανδικής Προεδρίας σας προς αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ ο Βόλκεν από Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ναι, καταρχάς να σας ευχαριστήσω. Έχω δύο ερωτήσεις ε, η πρώτη έχει να κάνει με τις αεροπορικές μεταφορές που σίγουρα είναι ο τομέας που αναπτύσσεται ταχύτερα σε ό,τι αφορά τις εκπομπές. Ε, και επίσης η κοινή γνώμη δίνει όλο και περισσότερη σημασία στο θέμα αυτό, πολύ περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα. Τι μέτρα λοιπόν εσείς θα θέλατε να προωθήσετε για να βρεθεί λύση. Δύο ε, πιθανότητες βλέπω ή να έχουμε ένα φόρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο την πρόταση αυτή δηλαδή ή ε, σε ό,τι αφορά τη, τα έσοδα από το ΦΠΑ και ε, σε πάλι εκεί ε, ευρωπαϊκό επίπεδο να βρεθούν κάποια μέτρα. Το δεύτερο τώρα μέχρι το 2021 μιλάει για 55% μείωση κύριε Φόντερ Λάιεν και καλό είναι αυτό σίγουρα, όμως είναι γρήγορα ιδίως έχοντας υπόψη ε, εθνικά δεσμευτικούς στόχους ε, ε, για το 2020 στο πλαίσιο του, της Συμφωνίας του Παρισιού. Πώς συνάδουν αυτά τα δύο. Uh, Martin Osik for Renew. Thank you, Chair. Uh, the Minister... Από το Renew. Κυρία Υπουργέ, σε ό,τι αφορά τη βιοποικιλότητα και την κυκλική οικονομία, χαίρομαι που είναι προτεραιότητε. Είμαι Σλοβάκο και χαίρομαι ιδιαίτερα που επίση και οι χώρε Κεντρική Ευρώπη μπορούν να αναδεσμευτούν στην ε, κλιματική ουδετερότητα προ τον άνθρακα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα τα εμπρό. Ποιο είναι το πρόβλημα όμω, Είναι ασυνεπεί μεταξύ του οι πολιτικέ. Ε, δηλαδή λέμε θα μειώσουμε τον άνθρακα από τη μία. Από την άλλη πλευρά είναι ένα ενωσιακό πρόβλημα το γεγονό ότι στηρίζουμε με στοχευμένες επιδοτήσεις και με εξαγωγές ε, πιστώσεων ή άλλα μέτρα τον τομέα αυτό. Άρα, τι θα κάνει η Φλαδική Προεδρία επ' αυτού. Και επίση, είναι ένα θέμα που δεν αναφέρατε αυτό. Δεν ξέρω αν θέλετε να το κλείσετε σε ό,τι αφορά την αξιονομία των πράσινων επενδύσεων. Θα το κλείσετε και αυτό το θέμα. Έλλη Μακέοντα από τους πράσινους. I... Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι από τη Σκοτία, που όπως και η Φιλανδία στηρίζει ναι. πιο φιλόδοξους κλιματικούς στόχους και αναγνωρίζει ότι επήγει το ζήτημα. Πρέπει λοιπόν όντως να τηρήσουμε την Συμφωνία των Παρισίων για να αποφύγουμε να ξεπεράσουμε την αύξηση των 1,5 βαθμού. Λοιπόν, πώς θα γίνει να εμείνουμε στις φιλοδοξίες μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα καθυστερεί όσον αφορά το στόχο της ε, κλιματικής ε, ε, ουδετερότητας, ουδετερότητας όσον αφορά το αποτύπωμα Μάθρακα. Τι θα δούμε στη Νέα Υόρκη, κυρίως με τις χώρες που έχουν ήδη πει ότι δεν θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο. Και ποιο θα είναι το βασικό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη διάσκεψη αυτή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για την Προεδρία σας. Μισελ Φιζίκ, ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Σλοβακικά, αν μου επιτρέπετε. Για να μπορέσουμε να έχουμε ουδετερότητα ως προς τον ανθρακά στο 2050, πρέπει να υλοποιήσουμε μια σειρά από μέτρα. Ποια είναι αυτά. Πώς θα εξασφαλίσουμε τη δέσμευση άνθρακα. Να την ε, περιορίσουμε σε σχέση με τις δυσμενείς συνθήκες που μπορεί να ε, φέρει στην δασοπονία. Ξέρουμε ότι η Φιλανδία έχει προχωρήσει ιδιαίτερα στην ε, βιοοικονομία, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην, στην ξυλία, στην μάζα από ξυλία αυτό δεν μπορεί να έχει όμως ε, συνέπειες για τα δάση και μάλιστα σε πολλά κράτη ευρωπαϊκά, στα οποία προσμετρώ και τη Σλοβακία, που έχουν ε, υποβάθμιση των δασών τους. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να παρασυρθούμε σε μια ε, απεριόριστη και αλόγιστη χρήση και κατάχρηση των δασών. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στου ομιλητέ, Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε, κυρία. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, κύριε Υπουργή, εμείς θέλουμε πολιτικές που να αντιμετωπίζει τις ανάγκες όλων. Η πρόκληση είναι να αλλάξουμε συνήθειες, να αλλάξουμε τρόπο ζωής, Υπάρχουν λοιπόν επιπτώσεις σε όλους τους τομείς, τον οικονομικό, τον κοινωνικό, το περιβαλλοντικό. Οι προκλήσεις δηλαδή είναι πολλέ και σε διάφορους τομείς. Η μετάβαση θα πρέπει να λάβει υπόψη τον κοινωνικό τομέα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μειώσουμε τις φιλοδοξίες μας. Όχι, πρέπει να τι καταστήσουμε δυνατόν εφικτέ και να φροντίσουμε για τους ε, ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται το θέμα της κλιματικής αλλαγής, αλλά κυρίως να ακούσουμε τους νέους, οι οποίοι διαμαρτύρονται και μιλούν για αυτή την κρίση όσον αφορά το περιβάλλον. Το θεματολόγιο του ΟΗΕ και οι βιώσιμοι στόχοι αποτελούν το κατάλληλο πλαίσιο. Συνεπώς, σας ζητώ δεδομένου ότι δεν υπάρχει στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα, πώς θα αντικατοπτρήσει τους βιώσιμους στόχου Ευρωπαϊκή Ένωση σε Φιλανδική Προεδρία και τις προσπάθειες των χωρών μελών στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, για παράδειγμα. Κατρίν Γκριζέ. Ταυτότητα και Δημοκρατία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, το κλίμα για σας θα είναι η πρώτη προτεραιότητα της Προεδρίας σας και είναι σημαντικό να έχουμε μια σωστή διάγνωση και στη συνέχεια να εφαρμόσουμε τα σωστά μέτρα. Οι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών που υπογράφουμε τη μία μετά την άλλη αυξάνουν τι εμπορικέ συναλλαγέ που ρηπαίνουν όλο και περισσότερο. Έτσι δεν σεβόμαστε του στόχου των Παρισιών. Κάποιες χώρες αποσύρονται εξάλλου, ενώ άλλες χώρες βάζουν στόχους που δεν είναι εφικτοί. Μιλάμε για 100 δισεκατομμύρια δολάρια που δίνουμε στις χώρες του Νότου και κάποιες από αυτές ε, χτίζουν καινούριε μονάδες άνθρακα, ενώ οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις εκφράσουν την ικανοποίησή τους. Τι άλλο θέλετε, η ιδεολογία αυτή των ελεύθερων συναλλαγών αντιβαίνει στην οικολογία. Μήπως, κυρία Υπουργέ, η λύση θα ήταν να σταματήσουμε αυτές τις μεγάλες παγκόσμιες συμφωνίες και να επιστρέψουμε στην τοπική κλίμακα, τα κράτη-μέλη να ελέγχουν τα σύνορά τους και να μπορούν έτσι να ανταποκριθούν καλύτερα στι ανάγκες τους. Πρόεδρος, ωραία, πέντε λεπτά παρακαλώ να επικεντρώσετε τις ερωτήσεις, απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Και έτσι να μπορέσουμε να αποκομίσουμε συγκεκριμένες προτάσεις ε, του Συμβουλίου και απαντήσεις του Συμβουλίου στις ανησυχίες μας. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας αυτές. Η πρώτη ερώτηση είχε να κάνει με την ανταγωνιστικότητα και ε, πώς αντιλαμβανόμαστε τις ε, διάφορες καταστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Όντως, η κυκλική οικονομία είναι ένας τρόπος να προχωρήσουμε και πρέπει να την προωθήσουμε. Θα βοηθήσει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά μας έτσι. Επίσης, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για το πώς θα περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή. Είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα, ένα συγκεκριμένο στόχος και θέλουμε να το φροντίσουμε κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας. Τώρα, ο κύριος Βίλκον μας ρώτησε για τις αεροπορικές μεταφορές. Αυτά είναι θέματα τα οποία εξετάζει το Συμβούλιο ε, Υπουργών Μεταφοράς. Ε, και ο κύριος Μάρτιν είναι σήμερα εδώ και συζητάει αυτό το θέμα με την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Η Φιλανδία θα οργανώσει πάντως μια επιπλέον συνάντηση των Υπουργών Μεταφοράς για να συζητηθεί ακριβώς αυτό το θέμα των στόχων, όχι μόνο για τις αεροπορικές μεταφορές, αλλά για παντός είδους μεταφορές. Πράγματι, χρειαζόμαστε αποφάσεις τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και τοπικά, για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τους στόχους και τις δεσμεύσεις μας ε, βάσει της Συμφωνίας των Παρισιών. Ξέρουμε ότι οι πολίτες μας θέλουν οικονομικά να μειώσουν τη ρήπανση από τις αεροπορικές μεταφορές. Τώρα πώς αυτό θα γίνει ακριβώς δεν ξέρω να σας το πω τώρα. Η επόμενη ερώτηση που μου τέθηκε είχε να κάνει με την βιώσιμη οικονομική ενίσχυση. Αυτό είναι θέμα των Υπουργών Οικονομικών. Η Υπουργός Λίμπηλα ασχολείται με αυτό το θέμα. Βέβαια και είναι σημαντικό να έχουμε βιώσιμα δημοσιονομικά και μια συμφωνία πάνω σε αυτό. Η Φιλανδική Προεδρία, πάντως, το έχει βάλει και αυτό στις προτεραιότητές της. Είναι πολύ σημαντικό για μας και ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε πάνω σε μια εντολή στο Συμβούλιο και να αρχίσουμε τον τριμερή διάλογο όσο γίνεται πιο γρήγορα, το φθινόπωρο. Η επόμενη ερώτηση ήταν της κυρίας Μακλίωτ, η οποία μας ρώτησε για την διάσκεψη του ΟΗΕ και ποια θα είναι η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, συζητήθηκε στο Άτυπο Συμβούλιο και είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογραμμίσει την δέσμευση που έχει αναλάβει στους ε, στόχους, μεταξύ άλλων και το στόχο του 1,5 βαθμού. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και πιο μακροχρόνιο στόχος πάνω στον οποίο πρέπει να δουλέψουμε στο Συμβούλιο. και είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό και το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υλοποιηθούν και θα συνεισφέρει σε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως πρέπει και οικονομικά. Αλλά είναι αλήθεια ότι παρόλο που έχουμε εξαιρετική νομοθεσία, οι χώρες μέλη είναι αυτές που πρέπει να δράσουν και να υλοποιήσουν αυτή την νομοθεσία. Αλλιώς δεν γίνεται. Έπειτα. Άλλη ερώτηση από τον κύριο Βίντσικ για τη χρήση γης και τα δάση. Φυσικά είναι κάτι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για την ε, κλιματική αλλαγή και τον περιορισμό της και πώς θα πετύχουμε τους στόχους των Παρισίων. Αλλά ακριβώ γι' αυτό πρέπει να κοιτάμε όχι μόνο τις εκπομπές, αλλά και τις ε, ε, λεκάνες που μας ε, δεσμεύουν το διοξίδιο του άνθρακα, όπως είναι τα δάση. Είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών, αλλά πρέπει να φροντίσουμε να υλοποιήσουμε την ε, οδηγία για την παράνομη ξυλία κλπ. Πράγματα πολύ σημαντικά. Είπαμε τα δάση όντως είναι πάρα πολύ σημαντικά σε σχέση με το κλίμα και την κλιματική αλλαγή. Ε, κυρία Μπουκάρτ τώρα, όσον αφορά τους βιώσιμους στόχους και την κλιματική μας πολιτική, είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας όλο τον κόσμο σε αυτό, σε αυτή την προσπάθεια. Μιλήσαμε πριν για τους νέους, οι οποίοι ανησυχούν όλος ιδιαίτερος και πρέπει να τους δώσουμε απαντήσεις πρέπει να φροντίσουμε κανένας να μην νιώθει ότι αυτός μόνο είναι που πληρώνει για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να υπάρχει κάποια ισότητα. Πολύ σημαντικό αυτό για την Προεδρία μας, να ξέρετε. Όπως επίσης, πολύ σημαντικό να ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί ότι τους έχουμε υπόψη μας όταν παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Η κυρία Γκριζέ τώρα με ρώτησε για τις εμπορικές συμφωνίες. Και πώς λαμβάνουμε υπόψη μας πώς τη λαμβάνουμε μας και πώς διασφαλίζουμε τους στόχους μας σε σχέση με τις εμπορικές αυτές συμφωνίες. Βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη φαντού. Δηλαδή, οι προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής να αποτελούν μέρος όλων των πολιτικών μας, όλων των κλάδων και όχι μόνο ενός. Αυτά. Σας ευχαριστώ και προχωρούμε στο τελευταίο γύρο ερωτήσεων. Επτά οι συνάδελφοι που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο, αλλά έχουν στήσει και άλλοι. Αν ε, μας δοθεί το περιθώριο, θα κοιτάξουμε βέβαια να προσθέσουμε και άλλους. Ξεκινώ λοιπόν. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πρώτο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ και ευχαριστώ που είστε εδώ. Είπατε ότι δεν θέλετε να συζητήσετε θέματα ιστορικής πολιτικής Φιλανδία. Ωστόσο φρονώ πως η πολιτική εμπειρία ενό πολιτικού από τη χώρα του ε, το ε, καθιστά και η θέση να αντιληφθεί και να αναλύσει και την ευρωπαϊκή πολιτική. Γι' αυτό με αυτό το πρίσμα θέλω να σας κάνω τις ερωτήσεις. Πρώτον λοιπόν, αλληλεξάρτηση στην παραγωγή της ενέργειας από τον άνθρακα. Θεωρείτε ότι το να περάσουμε από τον άνθρακα στη μαζική πυρηνική παραγωγή ενέργειας είναι κάτι το αποδεκτό, κάτι το θετικό καταρχάς για σας και κάτι το αποδεκτό για τον ε, Ευρωπαίο πολίτη εν γέννη. Δεύτερον, Θεωρείτε ότι μπορούμε να ξεφύγουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση από την μεγάλη εξάρτηση για τους υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία. Και κάτι ακόμη πάλι σχετικό με την εμπειρία σας από την Φιλανδία, αλλά όχι μόνο. Ναι, σας παρακαλώ πιο γρήγορα, λέει ο Πρόεδρος. Το μέλλον της χαλιβουργίας μέσα από την προοπτική των πολιτικών για το κλίμα, πώς το βλέπετε. Ευχαριστώ, Σε Βουενά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην ανάγκη καταπολέμησης της υπο... οικολογικής υποβάθμισης. Θα ξέρετε την υπόθεση της Ματρί Σεντράλ, μέτρα τα οποία έδωσαν πολύ καλά αποτελέσματα γιατί μείωσαν ε, τις εκπομπές οξυδίου του αζότου και ξέρετε ότι αυτό επηρεάζει τη ζωή και το επίπεδο διαβίωσης των ε, Μαδριλένων. Είχαμε πει επίσης ε, ότι δεν υπάρχει κατά της ακροδεξιάς ε, κορντών ε, ε, σανιτέρ. Δεν υπάρχει αποκλεισμό στη χώρα μας. Και το θέμα είναι τι μέτρα μπορούμε να προωθήσουμε που θα μειώνουν τι εκπόσει και θα βελτιώνουν το βετικό επίπεδο. Πρέπει να εκμεταλλευτείτε την Εξάμεινη Πρόεδρε, αν υπάρχουν μέτρα που βελτιώνουν τη δημόσια υγεία και μειώνουν τη ρήπανση στις πόλεις, να μην μπορούν να αναστραφούν, ε, να ανακληθούν τα μέτρα αυτά. Και σε ό,τι αφορά τα λίμματα για γεωργική χρήση, ε, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς προχωρούν αυτές οι συζητήσεις. Ε, σας το ζητώ, αν είναι δυνατόν, να βρεθεί, να δοθεί ένα αίσιο πέρα στις συζητήσεις αυτές. Ευχαριστώ. Thank uh, Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που είστε εδώ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η κλιματική αλλαγή και η κυκλική οικονομία είναι προτεραιότητες ε, της Προεδρίας σας. Και σχετικά ε, το ερώτημά μου είναι τι μέτρα θα προτείνετε για να το ότι η κυκλική οικονομία θα είναι ένα modus operandi σε όλους τους τομείς, ε, σε όλες τις αξιακές αλυσίδες, συγκεκριμένα ε, η σχέση μεταξύ κυκλικής οικονομίας και στόχων κλιματικής αλλαγής. Πώς θα τα συνδέσουμε αυτά και επειδή μιλήσατε για την Κομισιόν, έχει αξιολογηθεί η έκθεση με τα 54 μέτρα ε, δράσης ε, για την κυκλική οικονομία και ο τομέας της κλωστοϊφαντουργίας εντοπίζεται ως ένας από τους κλάδους πάνω στους οποίους χρειάζεται ακόμη δουλειά. Όπως γνωρίζετε, είναι εντατική χρήση πόρων, επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον ε, αυτή η βιομηχανία και έχει όμως και βαρύτητα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Τι σχέδια έχετε λοιπόν για να προωθήσετε το επίκεντρο στην κυκλική οικονομία στην κλωστοϊφαντουργία, λαμβάνοντα υπόψη ότι πρέπει να είμαστε συνεπείς προ προς τους στόχους για την κλιματική αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής Βιομηχανία. Ευχαριστώ και κάθε επιτυχία εύχομαι στην Προεδρία σα. E ε, Κυρία ECR. E ευχαριστώ πολύ. Και ξεκινώ ευχαριστώντας σας ε, για την παρουσία σας εδώ, για τη θεσμότητα να μιλήσουμε. Παρακολούθησα μεγάλο ενδιαφέρον την ε, τοποθέτησή σας και με ξεφνιάζει ιδιαίτερα το ότι βλέπω να εξισορροπείτε τις εκπομπές και τη μείωσή τους ή τον περιορισμό τους με χρονικό όριο του 2050 εκτός και αν μεταφράστηκαν λάθος τα λόγια σας. Κυρία Υπουργέ, Ε, οι μηχανίε στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες δυσκολίες και τα μέτρα για την κλιματική αλλαγή, το μόνο αποτέλεσμα που φέρνουν είναι να τις διώχνουν από την Ευρώπη και να τις στέλνουν σε άλλες χώρες. Και μάλιστα χώρες οι οποίες δεν τηρούν τους κλιματικούς στόχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνουν προϊόντα και τα αγοράζουμε από χώρες με πολύ ε, μεγάλο ίχνος διοξιδίου του άνθρακα. Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει η πολιτική μας να είναι τέτοια ώστε ε, να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας και την βιομηχανία μας. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για αυτά που είπατε για την ε, δίκαιη κοινωνικά μετατροπή των οικονομιών. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί αυτό. Βέβαια και η ενεργειακή φτώχεια είναι κάτι πολύ σημαντικό. Καλώς. Κοιτάξτε όμως σας διακόπτω, διότι δεν θα αφήσετε χρόνο στους λοιπούς συναδέλφους. Έχουμε ένα κανόνα και πρέπει να το τηρήσουμε. Κυρία Κόπα της Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που είστε εδώ. Διάβασα με προσοχή το πρόγραμμα της Προεδρίας σας. Ε, μπορώ να πω ότι συμφωνώ με τις προτεραιότητες σας στο σύνολό τους όπως τις περιγράφετε. Θα ήθελα ωστόσο να σταθώ στην ε, εξάρτηση από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής, για τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το κράτος δικαίου. Γιατί ναι, Βεβαίως και θέλω να διαφυλαχθεί η, κοινωνική, η κλιματική αλλαγή, να αντιμετωπιστεί μάλλον η κλιματική αλλαγή, αλλά να διαφυλαχθεί πάνω απ' όλα το κράτος δικαίου. Πώς λοιπόν θα γίνει αυτό χωρίς να ε, τεθούν σε κίνδυνο ε, μέτρα που χρειάζονται σε ορισμένα κράτη, για τα οποία όμως υπάρχει ο κίνδυνος να επιβληθούν κυρώσεις λόγω κράτους δικαίου. Γιατί να τιμωρήσουμε αυτούς τους πολίτες. Μήπω ο τρόπο θα ήταν να μην δίνουμε τα χρήματα κατευθείαν στι κυβερνήσει εκείνε οι οποίε παραβιάζουν το κράτο δικαίου, αλλά να πηγαίνουν τα κονδύλια ε, σε, στην τοπική αυτοδιοίκηση με κάποιο τρόπο να μην εξαρτώνται από τι κυβερνήσει, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ. Ακούσαμε από τα διάφορα στοιχεία που έχουμε ότι 3 δισεκατομμύρια δολάρια έφυγαν από τις χώρες τις ε, αναπτυγμένες χώρες τις αναπτυσσόμενες. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή με αυτό το σύστημα κεφαλαίου και της εξόριξης πόρων. Όσο παραμένει αυτό το σύστημα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τίποτα. Ε, δυστυχώς έχουμε τους φορολογικούς παραδείσους οι οποίοι φροντίζουν να μην μπορούν οι τοπικοί παράγοντες να φτιάξουν τις υποδομές που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές καταστροφές και αναγκάζει τον κόσμος να φεύγει από τα σπίτια του για να μπορέσει να επιζήσει. Κύριε Υπουργέ, πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έχουμε μια συνολική ολοκληρωμένη άποψη για το θέμα ή όχι και θα αντιταθείτε στη συμφωνία με τη Μερκοσούρ ναι ή όχι. Είναι καταστροφική για το περιβάλλον, θα επιδεινώσει την αποψήλωση των δασών γύρω από τον Αμαζόνιο και θα καταστρέψει και τους αγρότες οι οποίοι μπορούν να παράγουν καθαρά τρόφιμα που είναι κάτι που χρειάζεται η Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Μία γεγραμμένη. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ πέρα μιλάμε για ανταλλαγή απόψεων, για το κλίμα, για την βιοπικιλότητα. Οι Φιλανδοί είναι περήφανοι για τα δάση τους. Θέλω να μιλήσω εγώ τώρα για την αποψήλωση των δασών στην Κροατία. Την ε, διαφθορά την βλέπουμε στην Κροατία μέσω της αποψήλωσης των ε, δασών, γιατί πρόκειται για κρατικές επιχειρήσεις και τα σχέδια που γίνονται, μάλλον θα έπρεπε να γίνονται 100 χρόνια νωρίτερα. Στην Κροατία 5 εκατομμύρια ε, τετραγωνικά ε, φυτέψαμε και τα τέσσερα ε, καταστράφηκαν. Τώρα είμαστε στα 7,5 και 6 εκατομμύρια καταστρέφονται από την υλοκομεία. Βέβαια αυτά τα νούμερα δεν σημαίνουν τίποτα για πολλούς, γιατί μπορεί μεν να υπάρχει πληθωρισμός στις τιμές, αλλά όχι στην στον υπολογισμό του ξύλου από την υλοτομία. Κανονικά θα έπρεπε τα δάση να προστατεύονται από το κράτος, από την επιχείρηση που διαχειρίζεται τα δάση. Πώς θα βάλουμε τέλος σε αυτή την κατάσταση. Πρόεδρος, 7 λεπτά μένουν. 5 ομιλητές θα πάρω στο ΚΑΤΣΔΙ. Ξέρω ότι υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Και αρχίζουμε το ΕΛΚ. Ο κύριος που σας ζήτησε το λόγο, δεν είναι όμως εδώ. Μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ σας ποιος θα τον αντικαταστήσει. Τρεις ήταν ποιος. Ένας. Ωραία. Εσείς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι που σας βλέπω εδώ. Είμαι από την Σλοβενία εγώ και το περιβάλλον για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και σε εσά. Κυρίως η ύπεθρος που θέλουμε να προστατεύσουμε. Πολλοί άνθρωποι από την ύπεθρο στις χώρες μας ε, ταξιδεύουν στις πόλεις, ακόμα και πηγαίνουν να εγκατασταθούν στις πόλεις. Πράγμα που σημαίνει ότι οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αυξάνονται στις πόλεις. Όταν μιλάμε λοιπόν για την βιοπικιλότητα, εμείς πρέπει να την προστατεύσουμε. Αυτό όμως έχει ένα τίμημα. Και οι γεωργοί χάνουν έσοδα γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν εξίσου τις εκτάσεις που διαθέτουν. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, τι σκοπεύετε να κάνετε για να προστατεύσετε την ύπεθρό μας και σκοπεύετε να δώσετε κονδύλια προς αυτό το σκοπό. Ευχαριστούμε η Μαρία Ρενά. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μία μελέτη που έγινε από 3.500 Αμερικανούς οικονομολόγους που δείχνει ότι αν συμπεριλάβουμε στις εκπομπές ε, δεξιδίου του άνθρακα και την κατανάλωση, τότε ε, τα ποσά για την Ευρώπη θα ήταν αυξημένα κατά 30%. Η κυρία Φοντερ Λάιεν ήρθε με μία οριακή πρόταση ε, μάλλον ήρθε με μια πρόταση που έχει να κάνει με τον άνθρακα και τη φορολόγησή του στα σύνορα. Εσείς ως Προεδρία του Συμβουλίου θα προτείνετε ένα εργαλείο έτσι ώστε να αντιμετωπίσετε αυτά που λένε οι οικονομολόγοι και συγχρόνως να λάβετε υπόψη σας αυτά που προβλέπονται στις εμπορικές συμφωνίες. Νικόλα Στεφανούτα τώρα από το Ρινιού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ Μίκονεν, Έρχεται το καλοκαίρι, αλλά αυτό σημαίνει ότι έρχονται και ακραία καιρικά φαινόμενα. Κάθε χρόνο βλέπουμε ότι επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία. Στις χώρες μας, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, θα έρθουν διάφορες χώρες και θα ζητήσουν ε, χρήματα από το Ταμείο Αλληλεγγύης και λοιπόν, όπως και η χώρα μου η Ρουμανία, ε, είχε πρόσβαση 18 φορές. Δηλαδή, αντί να φροντίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που χρειάζονται για να αντιμετωπίζονται τέτοια φαινόμενα, αφού έχουν προκύψει ζητάμε εκτάκτως ε, βοήθεια. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχουν αρκετά χρήματα, αρκετοί πόροι για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις ε, κλιματικές κρίσεις, με τις οποίες κανείς από μόνος του, καμιά από τις χώρες μας από μόνη της, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Ε, κυρία Χωτάλα, εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση εγώ για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την αποψήλωση των δασών. Πώς θα αντιμετωπιστεί. Σήμερα θα δημοσιευθεί και όπως είπε και η κυρία Ρενά, πολλές από τις δικές μας εκπομπές ουσιαστικά είναι εισαγωγή, εισάγονται. Υπάρχει υπόσχεση να κοιτάξουμε τη δέωση επιμέλεια όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τις εκπομπές και πρέπει να το κάνουμε αυτό για να μην εισάγουμε τελικά εμείς κλιματική αλλαγή απ' Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, δεν θα ήταν κάτι που θα έπρεπε να εξετάσει και το Συμβούλιο Περιβάλλοντος και όχι μόνο εκείνο της Γεωργίας ή Δασόνη, δεν ξέρω τι, γιατί είναι συνολικό το θέμα, οπότε σας παρακαλώ βάλτε το και στους Υπουργούς Περιβάλλοντος το Συμβούλιο. Ευχαριστούμε. Τέλος, η κυρία Βελιούσκα από το ECR παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, κύριε Υπουργέ. Σας εύχομαι πάνω απ' όλα μεγάλη αποφασιστικότητα και επιμονή. Γιατί δεν έχετε εξάμεινο μπροστά σας, αλλά τρίμηνο. Και έχετε να συζητήσετε και το νέο προϋπολογισμό με μια νέα επιτροπή. Που θα συσταθεί το νωρίτερο στα τέλη Σεπτεμβρίου. Και ερώτηση. Έχετε καμιά ιδέα για το πώς πρέπει να διαμορφωθεί ο προϋπολογισμός, τι επίπεδα θα έχει και πάνω απ' όλα τι θα περιλαμβάνει ως προς την προστασία των υδάτων, εάν θα υπάρχουν κάποιες πρόνοιες. Όταν μιλούμε για κυκλική χρήση των ε, νερών, κυκλική οικονομία, δεν μιλούμε μόνο για το νερό, αλλά και για την ανακύκληση και ε, επισκευή και νέα χρήση των αντικειμένων. Παρακαλώ, υπουργό για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ο πρώτος ε, μίλησε για την ε, παραγωγή ενέργειας και τι λύσεις υπάρχουν. Ποιε είναι οι φιλανδικέ εμπειρίε και οι φιλανδικέ λύσει. Θα ήμουν ευτυχή να τα συζητήσουμε. Αλλά δεν μιλώ εξ ονόματος της χώρας μου αυτή τη στιγμή, μιλώ εξ ονόματος του Συμβουλίου συνολικά. Σίγουρα το μέσο τη ενέργεια έχει να διαδραματίσει ένα κρίσιμο ρόλο για την επίτευξη των κλιματικών στόχων. Αυτό αφορά όλε τι χώρε. Και σημαίνει ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να έχουμε μια πιο σύντομη χρονικά μετάβαση. Και αν δείτε ποιες είναι οι φιλανδικές λύσεις, δεν θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν πυρηνική ενέργεια. Επαναχρησιμοποίηση του νερού, των λιμάτων συγκεκριμένα, τον κύριο Λουενά Νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση και θα εγκριθεί η επιφυλακτική προεδρία ο σχετικό κανονισμό και ο στόχο αυτό είναι σημαντικό. Σόλι Πέρε. Ζήτησε απτές δράσεις για την κυκλική οικονομία. Η κυκλική οικονομία σίγουρα αποτελεί προτεραιότητα της Φιλανδίας. Σίγουρα θέλουμε να περιορίσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Μιλήσατε για την φαντουργία. Πράγματι, είναι ένας τομέας τον οποίο πρέπει να δούμε εκ του Σίγουρα η φαντουργία προσφέρει πολλές ευκαιρίες και μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους μας με πολύ πιο αηφόρο τρόπο. Για να είναι λιγότερος ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος αυτού του κλάδου. Σε ό,τι αφορά τώρα την κυρία Βυσνιεύσκα. Σε ό,τι αφορά την δίκαιη μετάβαση. Μιλήσατε για τις διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ε, οι διαφορετικές για να πετύχουν ουδετερότητες προς τον άνθρακα. Η Φιλανδία σίγουρα θέλει να γίνουν συζητήσεις με τα κράτη-μέλη. Και σίγουρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι διαφορετικές οι αφετηρίες, αλλά ο στόχος είναι σημαντικός και κοινός. Κόβατς. κράτος δικαίου. Πράγματι είναι πολύ σημαντικό ε, αυτό το θέμα. Δεν είναι όμως το δικό μου χαρτοφυλάκι, άρα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Απλά σας λέω ότι είναι προτεραιότητά μας και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Wallis. Μίλησατε για τη συμφωνία με τις χώρες Μερκοσούρ. Σίγουρα υπάρχουν λόγια ανησυχία, αλλά νομίζω το συζητήσατε με τον Υπουργό Λέπα που είχε έρθει χθε στην Επιτροπή σας. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η συμφωνία να περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σίγουρα πρέπει να τα δούμε διαφορετικά τα πράγματα και η αρχή της προφύλαξης είναι μια αρχή που πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνεται όταν τίθεται θέμα λήψης αποφάσεων με περιβαλλοντικό αντίκτυπο για την Χάιντι Χάουταλα. Μιλήσατε για την αποψήλωση των δασών, που είναι πραγματικά ένα σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποψήλωση που επίκειται από ό,τι ξέρετε. Μιλά βέβαια συνολικά για το θέμα αυτό και ζητείται βελτίωση με την καλύτερη αξιοποίηση των εφιστάμενων εργαλείων και μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώ. Η Φιλανδία είναι έτοιμη και διτεθειμένη να καταπολεμήσει το πρόβλημα της αποψήλωση των δασών και στο πλαίσιο της Προεδρίας μας. Όταν δε δημοσιοποιηθεί αυτή η ανακοίνωση της Κομισιόν θα τη μελετήσουμε και θα την εξετάσουμε από το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής και της βιοπικιλότητας. Υπήρχε και ένα άλλο ερώτημα, το οποίο, για να δω, πώς θα εξασφαλίσουμε μια ευρύτερη, μια παγκόσμια συμμετοχή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πώς μπορούν και οι εμπορικές συμφωνίες να παίξουν ένα ρόλο. Φυσικά και πρέπει να συνεργαστούμε, διότι οι περισσότερες εκπομπές άνθρακα προέρχονται από την κατανάλωση εμπορευμάτων, αγαθών, τα οποία παράγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά και πρέπει να κάνουμε πάντα δυνατόν για να συνυπολογίζεται ο κλιματικός αντίκτυπος, περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο και πρέπει σίγουρα να βελτιωθούν τα καταναλωτικά πρότυπα, οι καταναλωτικές συνήθειες. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων Για σήμερα το πρωί θέλω να ευχαριστήσω την Υπουργό. Τηρήσαμε το χρονοδιάγραμμα, θα κάνουμε λίγα λεπτά διάλειμμα και μετά θα προχωρήσουμε στη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων με αρμόδια για τα θέματα κοινωνικών οικογενειακά ζητήματα. Σε πέντε λεπτά θα συνεχίσουμε.